Um, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ορίσατε στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής μας εδώ στο Στρασβούργο. Είδατε την ε, προτινόμενη μισή διάταξη για την απόψη μας συνεδρίαση. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες. και ηλεκτρονικά διατίθεται ο φάκελος στο application. Επίσης έχουμε και ζωντανή αναμετάδοση τη συνεδρίασής μας στο διαδίκτυο. Θέλω να σας ενημερώσω για μια άτυπη συνάντηση με την κυρία Άινη, που είναι η πρόεδρος του Συνασπισμού Φιλοδοξιών και πρόεδρο της Δημοκρατίας των Ίσων Μάρσαλ. επισκέπτεται η Πρόεδρος ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συζήτηση της Ολομέλειας σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων και εκεί εντάχθηκε και αυτή η συνάντηση που θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πάρα πολύ υποκοδομητική συζήτηση με την ηγέτηδα μιας από τις χώρες που θα πληγούν περισσότερο από αυτές τις εξελίξεις εν και της 23ης ε, κόπτο Νοέμβριο. Θέλω να είστε πολυπληθής στην συνεδρίαση αυτή που θα λάβει η χώρα από τις 9 έως 10 και μισή περίπου την Τετάρτη το πρωί. Τετάρτη, 14 Τετάρτη Ιουνίου. Ποιος είναι ο βασικός λόγος τώρα αυτής της ε, συνεδρίασης που έχουμε σήμερα είναι να ακούσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον ε, κύριο Τίμερμανς τον οποίο θέλω να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Κύριε να χαίρεστε πολύ σίγουρα που βρίσκεστε εδώ, γιατί και εμείς παρακολουθούμε τους του σύνεγγυς τις δραστηριότητές σας, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσετε να πραγματοποιηθούν οι ιδέες μας και οι ελπίδες μας για το μέλλον. Να ξέρετε ότι τα θέματα που σχετίζονται με το κλίμα είναι προτεραιότητα μεταξύ άλλων στην Επιτροπή μας και θα παραμείνουν ύψη στην προτεραιότητα μέχρι τα τέλη της ε, νομοθετικής περίοδου. Γνωρίζετε ότι έχουμε έναν τεμερή διάλογο για το ETS, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Έχουμε άλλα θέματα όπως ο Υπνισμός Προσπαθειών, το LULUCF, το πακέτο μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Και γενικώ θεωρούμε ότι με τα πακέτα μπορούμε να επικοινωνούμε με την κοινή γνώμη. Βέβαια έχουμε και πολυφαρτωμένο πρόγραμμα και έργο να επιτελέσουμε, αλλά είμαστε ευγνώμονες για αυτές τις προτάσεις. Τώρα, φερόντας τις δικές σας οριζόντιες ευθύνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Είμαι βεβαία και γνωρίζω ότι και εσάς σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να συνοθεί πρόοδος. Θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερα για τη γενική προσέγγιση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα και ιδιαίτερα θα μας ενδιαφέρει να μας πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας για την υλοποίηση των στόχων ε, της βιώσιμης ανάπτυξης ό,τι αφορά τις και εξωτερικές πολιτικές της Ένωση. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή η ΕΝΒΙ επεξεργάζεται μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία για τη δράση τη Ένωση για την ε, βιωσιμότητα. Επίση, απεστάλλει πρόσφατα και μια αντιπροσωπεία μα την ε, διάσκεψη για του ωκεανού, σε ό,τι αφορά τον 14ο αναπτυξιακό στόχο τη χιλιετία. Θέλουμε επίση να μα πείτε πώ σχεδιάζετε να υλοποιήσετε το σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία και να μα μιλήσετε ιδίω εφόσον αυτό είναι δυνατό, για τη στρατηγική σε σχέση με τα πλαστικά που μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω ε, άλλο, αλλά να πω κάτι ακόμη. Τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων είναι πολύ σημαντικά. Το είπα και στη συνάντηση ΣΥΣΥΣΥ. Δεν μας ικανοποιεί πρόοδος που έχει επιτελεστεί μέχρι στιγμής, ιδίως ό,τι αφορά την ε, αντοχή στα αντιβιωτικά. Διότι Είχαμε ζητήσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επανειλημμένως μάλιστα να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης που θα έρθει ως συνέχεια το σχέδιο δράσης που εξέπνευσε την προηγούμενη χρονιά. Και ελπίζαμε να συνοδεύεται και από νομοθετικά μέτρα αυτό το σχέδιο δράσης. Συν το ότι ακόμα περιμένουμε η Κομισιόν να σημειώσει πρόοδο και σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων ε, για τα κτηνιατρικά φάρμακα που έχει κολλήσει στο επίπεδο του Συμβουλίου αλλά είναι κάτι άκρος επίκαιρο και αναγκαίο. Να καλωσορίσω για μια ακόμη φορά του αδέλφους και κύριε Πρόεδρε, είστε ευπρόσδεκτο. Χαίρομαι που είστε εδώ και παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση για την προετοιμασία του προσεχούς προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να ακούσω τις απόψεις των μελών της Επιτροπής σας που είναι μια από τις σημαντικότερες επιτροπές για την κοινή ε, διακήρυξη ότι αφορά τις νομοθετικές προτεραιότητες και για φέτο ξέρω ότι εργάζεστε εντατικά πάνω σε τέσσερις προτάσεις ε, για τη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα, απορρίμματα και τρεις ε, νομοθετικούς φακέλους για τα συστήματα εμπορίας εκπομπών. Επίσης ασχολείστε και με τα θέματα της καθαρής ενέργειας για όλους. Καταρχάς θα ήθελα να, αναφέρω στο να αναφερθώ στο θεματολόγιο που καθοδηγεί και δίνει όραμα και στόχο τη δράση μας, που είναι το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους ε, στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Εγώ προσωπικά και οι Κομισιόν συνολικά έχουμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση και την παίρνουμε πολύ σοβαρά και εντό Ένωση και σε σχέση με τη συνεργασία που έχουμε με τι τρίτε χώρε. Ε, οι 17 στόχοι τη βιώσιμη ε, ανάπτυξη ε, είναι πολύ σημαντικοί για να βάλουμε του περιβαλλοντικού στόχου στο επίκεντρο του παγκόσμιου θεματολογία. Πέρσι τον Νοέμβριο Παρουσιάσαμε την ε, αντίδρασή μα στο Θεματολόγιο του 2030 και στόχου ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη και περιμένω να, ακούσω και τη, να διαβάσω και τη δική σα έκθεση σε σχέση με τη δική μα ανακοίνωση. Στόχο είναι να διατηρήσουμε την ορμή και όλα αυτά να τα μεταφράσουμε σε συγκεκριμένε πολιτικέ ε, και να λάβουμε σχετικέ αποφάσει σε παγκόσμιο περιφερειακό εθνικό επίπεδο. Η απάντησή μα ό,τι αφορά το Θεματολόγιο του 30 θα περιλαμβάνει δύο βασικού άξονε. Πρώτο άξονα είναι να ξορθολογήσουμε και να περιλάβουμε στο πλαίσιο πολιτικών και σε όλες τις προτεραιότητές μας τους βιώσιμους αυτούς στόχους, ιδίω ό,τι αφορά και τον προβληματισμό που πρέπει να ξεκινήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη της, του μακροπρόθεσμου οράματος. Και επίσης ε, θέλουμε να εστιάσουμε σε τομεακές πολιτικές ε, και στο όραμα αυτό μετά το 2020. Βασικός μας στόχος σίγουρα είναι να, να δούμε πώς θα πετύχουμε τους στόχους του 2020, αλλά αυτό που θα κάνουμε μέχρι το 2020 θα πρέπει να συνάδει και με το θεματολόγιο που θα μας φέρει στο 2030. Αυτή είναι η πιστεύω λογική συμβίωση των δύο αυτών αξών. Θέλουμε να αναπτύξουμε το μακροπρόθεσμο αυτό όραμα σε στενή συνεργασία με την πλατφόρμα των ενδιαφερομένων μερών που έχουμε δρομολογήσει, αλλά και από με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι θα είναι κρίσιμο ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τη δημιουργία πολιτικών και ρυθμιστικών πλαισίων που θα ενθαρρύνουν κυβερνήσει, πολίτε, επιχειρήσει να στηρίξουν ε, την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση για όλου. Κάτι που είναι απαιτούμενο, θέλουμε να πετύχουμε του στόχους Τη βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι το κοινό μα όραμα για τον κόσμο και έχοντα υπόψη τι πρόσφατε πολύ ατυχεί αποφάσει τη κυβέρνηση των ΗΠΑ για να, αποχώρησή του από τη Συμφωνία των Παρισίων είναι πάρα πολύ σημαντικό Εμεί στην Ευρώπη να παραμείνουμε όσο δυνατόν πιο ενωμένοι και προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο και να δείξουμε ε, ηγετική ε, προσέγγιση. Είναι μεγάλη πρόκληση και πρέπει να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξη και κοινωνικής ασφάλειας και προστασία. Θέλουμε ένα ισχυρό κοινωνικό συμβόλαιο. Ταυτόχρονα όμω, θέλουμε να μειώσουμε και το φόρτο και το βάρο στου φυσικού πόρου ε, και στον πλανήτη μα. Θα αυξηθούν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες περιοχές και θα πάρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι των φυσικών πόρων. Θα πρέπει εμεί λοιπόν να του δείξουμε ε, το σωστό παράδειγμα ότι μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία με ψηλά επίπεδα προστασία, αλλά με μειωμένο φόρτο σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Άρα σημαντικό παράδειγμα είναι και το πακέτο για την κυκλική οικονομία. Γιατί μπορεί αυτό να συνεισφέρει στη μείωση των απορριμμάτων, αποβλήτων, πλαστικών, θαλάσσιων αποβλήτων, ε, να περιορίσει την σπάνιδα του νερού, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πόρων και να δημιουργήσει θέσει εργασία και ανάπτυξη. Και το πακέτο για τα απόβλητα, για τα πάνω, είναι σημαντικό κομμάτι τη κυκλική οικονομία. Είναι προτεραιότητα και για, τους, ε, για τα τρία θεσμικά όργανα και θέλουμε να πετύχουμε γρήγορα πρόοδο. Να έχουμε μια συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτου και βασίζομαι και στη φιλοδοξία και τη σκληρή δουλειά τη δική σα τώρα που έχουν ξεκινήσει και τρεμερεί διάλογοι. Η διαχείριση των φοιτών με τον ε, σωστό τρόπο είναι κάτι που θα έχει μόνο κερδισμένου και μιλάμε εδώ για οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία εργασία, καινοτομία και για το περιβάλλον και για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν θέλει να διατηρήσει μεγάλη φιλοδοξία για το συνολικό πακέτο με βάση φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση και τη μείωση των οματερών αλλά και για ε, δίκαιους, ε, σωστούς, διαφανείς κανόνες υπολογισμού. Πρέπει να είμαστε στο ίδιο επίπεδο, να είμαστε στο ίδιο μικρό για να μπορούμε να συγκρίνουμε τι κάνουμε στα διάφορα κράτη-μέλη. Ίσως χρειαστεί ε, περισσότερος χρόνο για την επίτευξη των στόχων σε κάποιες χώρες. Υπάρχει συμφωνία από αυτού, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις ε, ακριβώς λόγω του επίπεδου της φιλοδοξίας μας. Ίσως θα πρέπει να συνοδευτεί αυτό από μεγαλύτερη υποστήριξη, όχι όμως με αναβολές. Ε, και οι προτάσει αυτέ είναι φιλόδοξε και σε ό,τι αφορά τα επίπεδα των στόχων, αλλά και σε ό,τι αφορά του κανόνε υπολογισμού. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Και είναι θετικό το ότι και Κοινοβούλιο και Συμβούλιο επιθυμούν να πετύχουν το μεγαλύτερο βαθμό συγκρισιμότητα και ισότιμο πεδίο ε, μεταξύ των κρατών μελών. Οι κανόνες υπολογισμού για την ανακύκλωση και τις χωματές θα πρέπει να είναι στέρεοι και πρακτικοί και διαφανείς. Επίσης, θέλουμε να προωθήσουμε την ιεραρχία των απολύτων και να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους με μια ευρύτερη καλύτερη χρήση οικονομικών εργαλείων όπως τη μεγαλύτερη ευθύνη του παραγωγού, του κατασκευαστή. Επίσης αναγνωρίζουμε τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για νέους ποσοτικούς στόχους. Γενικώ όμως αυτό το έργο θα πρέπει να καθοδηγείται από συνεκτικά αξιόπιστα δεδομένα και μία εκ των προτέρων ε, μελέτη αντικτύπου. Θα μελετήσω ιδιαίτερα το θέμα των ε, τροφικών αποβλήτων τροφίμων. Ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει την πρωτοβουλία της Πράσινης Κάρτας και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε. Επίσης υπάρχουν και πολλές άλλες πρωτοβουλίες ε, που θα ήθελαν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να αναλάβουμε εμείς ε, στον τομέα των αποβλητών και θα τα συζητήσουμε και με εσά και με τους συναδέλφους μου. Επίσης ε, περιμένουμε να έχουμε επικοδομητική συνεργασία με τους δύο νομοθέτες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τη διαδικασία και να έχουμε μια φιλόδοξη γρήγορη συμφωνία. Και επειδή το είπατε και εσεί, Πρόεδρε, τώρα θέλω να αναφέρω κάτι επίση σημαντικό στο πλαίσιο τη κεντρά για την οικονομία, που είναι τα πλαστικά. Γνωρίζουμε το πλαστικό ε, έχει σημαντικό χώρο στην καθημερινότητά μας, στις οικονομίες μας, αλλά ξέρουμε και ότι έχει και πάρα πολύ αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις. Το 70% σχεδόν των πλαστικών αποβλήτων είτε καίγεται, αποτεφρώνεται είτε κατέληξε σε 5 με 13 εκατομμύρια τόνοι κατέληξε στο περιβάλλον κάθε χρόνο, δημιουργώντας ωκεανούς πλαστικών αποβλήτων. Και αυτό είναι επιβλαβές για τη φύση, την οικονομία και την υγεία μας. Και στην Ολλανδία αποδείχθηκε πρόσφατα ότι αυτά τα πόματα ε, που μπορεί να είναι βιοδιασπόμενα, τα ε, μπουκάλια, αλλά τα ε, πόματα δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και κυρίως και στη θάλασσα. Πολύ δουλειά έχουμε να κάνουμε σήμερα. Πάνω από 1% του πλαστικού παράγεται από παρθένο υλικό και έχουμε 400 περίπου εκατομμύρια τόνους ε, θερμοκυπριακών αερίων ε, συνολικά το χρόνο από την παραγωγή πλαστικού. Και αν συνεχιστεί έτσι, μέχρι το 2050 θα έχουμε 15% ε, των παγκόσμιων εκπομπών ε, διοξείδιο το πλαστικό, πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Να δούμε που θέλουμε να είμαστε 10-20 χρόνια. Θέλουμε να δούμε λοιπόν το συνολικό κύκλο ζωή του υλικού αυτού και το πρώτο που παράγει από το πλαστικό. Γι' αυτό λαμβάνουμε μέτρα για να εφαρμόσουμε τι εφιστάμενε απαιτήσει. Ξέρετε ότι περιλαμβάνεται ε, η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στις νομοθετικές μας προτάσεις και το eco design θα το προωθήσουμε, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα με τα πλαστικά. Και γι' αυτό μέχρι τα τέλη του έτους θα δημοσιεύσουμε και μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το πλαστικό που θα ξεκινήσει τη διαδικασία άρδινα μετασχηματισμού της μελέτης, παραγωγής, χρήσης, διαχείρισης ε, του πλαστικού στο τέλος του κύκλου ζωής. Και θα δημιουργήσει τα θεμέλια για μια νέα βιομηχανία πλαστικού να είναι πλήρως κυκλική αυτή ε, η, βιομηχανία. Και αν αξιοποιήσουμε την όθηση και τα πετύχουμε αυτά, τότε όχι μόνο θα λύσουμε τέρας τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, θα αποκτήσουμε και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο προσκήνιο, δημιουργώντα πολλέ αναπτυξικέ ευκαιρίε στην Ευρώπη. Σε στρατηγική θα φαίνονται λοιπόν ποιε είναι οι φιλοδοξίες μας. Θέλουμε να αποσυνδέσουμε την παραγωγή πλαστικού από τη χρήση μη ανανόσιμων πόρων. Θέλουμε τα πλαστικά προϊόντα να είναι αποδοτικά, να μπορούν να κυκλώνονται και το αποτύπωμα άθρακα, ε, επίπτωση να είναι χαμηλή, μεγάλη να είναι η αντοχή και να μην έχουμε ε, πλαστικά απόβλητα που να μολύνουν το περιβάλλον. Τα μικροπλαστικά είναι μια πρόκληση πολύ σοβαρή και πολλοί διεθνεί φορεί όπω και είπα έχουν ε, πάρει μέτρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Πολλοί απαγορεύουν δουλεύουν τα μικροπλαστικά σε διάφορα προϊόντα και οι ερευνητέ αναπτύσσουν περιβαλλοντικά βιώσιμε εναλλακτικέ. Η στρατηγική θα αντιμετωπίσει και τα διασπόμενα πλαστικά. Μπορεί με, να φέρω ότι θα μπορούσε αυτό να είναι μια λύση για τη μείωση τη διαρροή του πλαστικού στο περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να είναι βιώσιμα και αυτά τα υλικά για την προετοιμασία στρατηγική, ότι οργανώνουμε στοχευμένε διαβουλεύσει με του δικομένου φορεί και θα έχουμε και μια συνεδρίαση, μια διάσκεψη όλων αυτών στι 26 Σεπτεμβρίου. Και τέλο, να πω δύο λόγια για τις μεθόδους εργασίας μας. Ε, αντίθετα με κάποιους, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αντίφαση μεταξύ καλύτερης νομοθεσίας αφενό και υψηλών περιβαλλοντικών πρότυπων αυτών. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο, γιατί η καλύτερη νομοθεσία δεν είναι μόνο πώς θα πετύχουμε του στόχου μα ε, απλά, ε, αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχουμε τι στόχους μας ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε ένα σχέδιο δράσης για την ε, περιβαλλοντική υποβολή αναφορών. Είχαμε κάνει ένα check-up όλων των διαδικασιών υποβολή αναφορών. Θέλουμε να έχουμε ποιοτικότερε πληροφορίε που θα παρέχονται πιο εύκολα και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρύτερα και αυτό θα ωφελήσει όλου όσου ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Και είχαμε και ένα πρόσφατο check-up των οδηγιών για τα πτηνά και τα οικοσυστήματα. Και είδαμε ότι ναι, μεν είναι κατάλληλε αυτέ οι οδηγίε για την έκπληξη του σκοπού του, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθούν καλύτερα για να είναι πιο αποτελεσματικέ οι οδηγίε. Και ακόμη όταν δεν χρειάστηκε με τι εξολογήσει μα να προτείνουμε νομοθετικέ αλλαγέ, παρόλα αυτά καταφέραμε να συζητήσουμε με του ε, εμπλεκόμενε φορεί να καταλάβουμε καλύτερα τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε για κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά, παραδείγματο χάρη, για τα πτηνά και τα οικοσυστήματα, με τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ πλέον έχουμε πολύ στενότερη συνεργασία που ήταν και οι αρχέ παραπώνουν το περισσότερο για αυτή τη διαδικασία, τι οδηγίε. Και θέλουμε με αυτή την αλληλεπίδραση να τα υλοποιήσουμε πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Υπερεύει λίγο ε, το χρόνο που μου είχατε δώσει και τώρα βέβαια προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Είπατε, μιλήσατε για τη σημασία του πακέτου για τα απόβλητα. Έχουμε εδώ τον εισηγητή. Έχουμε ξεκινήσει τον τριμερή διάλογο και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο Βέλα που στηρίζει την άποψη του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο. Στόχο είναι βέβαια να προωθήσουμε την καλύτερη δυνατή πολιτική και χαίρομαι για αυτό που είπατε, ότι χρειαζόμαστε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και πρέπει να τους εντάξουμε στο συνολικό πλαίσιο πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλώντας για την βέλτιστη ε, νομοθέτηση, ε, παρατηρούμε τις προσπάθειές σας ε, μέσω της διαδικασίας του Omnibus, όμως θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις προθέσεις σας σε ό,τι αφορά τη διαγραφή κάποιων διαδικασιών που επιβαρύνουν προκειμένου να σας υποστηρίξουμε. Παρακαλώ πολύ δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, όμως έχουμε και διάφορους συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές και κυρίως με τον κύριο Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο τη Κομισιόν για τι αοκέ του παρατηρήσει ε, και στηρίζω ιδιαίτερα αυτό που είπατε για τα πλαστικά. Και θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί αν είχαμε την πρόταση και τη Κομισιόν για τη στρατηγική ε, για τα πλαστικά. Ε, όμως θέλω να πω αυτό που είπε και η κυρία Βαλεάν, ε, last but not least. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία. Και δεν ξέρω αν έχω αντιληφθεί σωστά τα πράγματα, αλλά ναι. Και από εσάς και από τον ε, κύριο Γιούνκερ δεν έχω ακούσει μια πρόταση για το θέμα της υγείας ε, και πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ε, επικριτικά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να κάνουμε κάτι, παραδείγματο χάρη για τα αντιβιωτικά, την αντοχή στα αντιβιωτικά. Αυτό το αναφέρατε αλλά θα ήθελα να ε, πω ότι έχουμε και μια πρόταση της Κομισιόν, ε, την οποία έχουμε χαρακτηρίσει ευπρόσδεκτη, αλλά θα πρέπει αν έχουμε ε, νέα αντιβιωτικά για τα ζώα, κτηνιατρικά φάρμακα, έχουμε κάποια κίνητρα. Τι γίνεται όμως για την παρασκευή νέων αντιβιωτικών για τον άνθρωπο. και δεν έχει κάνει κάποια πρόταση η Κομισιόν. Θέλουμε να μετριάσουμε την αντοχή στα αντιβιωτικά ε, και την αντικροβιακή αντοχή. Θα πρέπει λοιπόν ε, να στηριχτούν οι προσπάθειες ε, μεν για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, δεν θέλω επειδή δεν έχουμε χρόνο να τα αναφέρω τώρα διεξοδικά, αλλά και στις συνθήκες λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα για τα θέματα της υγείας, όχι αποκλειστική βέβαια, Υπάρχει όμως αρμοδιότητα, υπάρχουν νομικές βάσεις, υπάρχουν δυνατότητες ε, και αν ε, ρωτήσει κανείς τους πολίτες ε, την ημέρα των γενεθλίων τους ή τη νέα χρονιά τι θέλατε, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οικονομική ανάπτυξη, όχι, αυτό που λένε όλοι η υγεία. Η υγεία είναι το πάνω, υγεία είναι το πρώτο. πρέπει λοιπόν να δώσουμε και εμεί σωστέ απαντήσει σε αυτό και ότι έχουμε ευθύνη. Ευχαριστώ. Και εγώ κύριε Λίζε. Ε, τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που μας υπογραμμίσατε τις προτεραιότητες σας. Τις μοιραζόμαστε και εμείς. Θα ήθελα να εστιάσω σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αναφέρατε. Την γλυφοσάτη συγκεκριμένα, το οποίο έχει γίνει θέμα πολιτικής ε, σημασίας από τότε που, ε, που ενδεχομένως υπάρχουν ενδείξεις ε, καρκινογένεσης αλλά και, αντε... και αντίθετες ενδείξεις. Ε, οι επιστημονικές ε, έρευνες αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής για να χαρακτηρίσουν την αρτηριστή γλυφασάτη ε, ως επικίνδυνη ουσία. Έτσι λέτε ως Κομισιόν. Εσείς ε, ως υπεύθυνος για την διαδικασία REFIT μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με την αξιολόγηση REFIT για τον κανονισμό για τα, ε, για τα νέα προϊόντα και τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία σκοπεύει να λάβει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά την διαφάνεια και την ε, επιστημονική αξιολόγηση από ομοτήμους για δραστικές ουσίες. Επίσης για το ίδιο θέμα και η ΕΦΣΑ και η ΕΚΑ ε, έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι η ε, η ουσία αυτή δεν είναι ε, καταφανώς, ε, ε, δεν έχει καταφανώς καρκινογενή αποτελέσματα, δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία τους. Ευχαριστούμε κυρία Αντάλη. Ε, από το ECR δεν υπάρχει εκπρόσωπος. Η κυρία Βέρντερ για τους φιλελεύθερους. Θα ήθελα να δείξω δύο ζητήματα, εν συντομία. Πρώτον για τη στρατηγική βιοπικιλότητα και δεύτερον για το περιβαλλοντικό dumping. Μιλήσατε για το φυσικό περιβάλλον, αλλά η στρατηγική βιοπικιλότητα που έχει ως στόχο το 2020 ε, δεν καταλαβαίνουμε ποια μέτρα προβλέπετε, προβλέπει. Πώς μετρά τη βιοπικιλότητα η Κομισιόν. Ε, έχουμε πετύχει τους στόχους μας, τον τελευταίο σίγουρα όχι. Ε, γιατί αυτό που λένε οι παραγωγικές οργανώσεις συνεχώς και παντού είναι ότι η βιοπικιλότητα χάνεται με μεγάλους ρυθμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καταστροφικούς ρυθμούς. Δεύτερον, για το περιβαλλοντικό dumping. Ε, συζητάμε το Brexit και όσοι δεν το γνωρίζουν να σε ενημερωθούν ότι το, η Βρετανία έχει πρέον έναν καινούριο Υπουργό Περιβάλλοντος υπέρμαχο του Brexit ε, θα ήθελε να καταργήσει πλήρως ε, την νομοθεσία του περιβάλλον και όταν ήταν υπουργό Παιδείας ήθελε να βγάλει από το ορολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τα της κλιματικής αλλαγής. Οπότε οτιδήποτε και αν γίνει ε, με την Βρετανική κυβέρνηση ελπίζω ότι θα διασφαλίσετε πως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, δεν θα οδηγηθεί στην ατραπό του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ. Ε, και δεν θα προσπαθήσει να διαφύγει ε, τη περιβαλλοντική νομοθεσία, που κάτι που θα επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιο ο Τραμπ αρνείται το φαινόμενο τη κλιματική αλλαγή και ε, ε, απέστειλε τι από τη Συμφωνία των Παρισίων. Ε, θέλουμε να μην αποτελέσει μοντέλο και να μην μας μεταδώσει ε, περιβαλλοντικό ντάμπινγκ ε, στη δική μας περιοχή, εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Μπιάτα. Από, από την ΚΟΕ, η κυρία Κονέτσμα. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπατε ε, εσείς, αν μπορώ να το συνοψίσω. Εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Έχουμε όλο ένα και περισσότερη νομοθέτηση, αλλά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό που διαθέτουμε δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή στα κράτη-μέλη και παρόλα αυτά προετοιμάζουμε άλλα νομοθετήματα, ολοένα και περισσότερα. Αν όμως κάτι δεν εφαρμόζεται, δεν έχει νόημα να νομοθετούμε εκ νέου. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, κύριε Αντιπρόεδρε γιατί θα πρέπει να δούμε καταρχήν τη μη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Εσείς έχετε ε, ανταποκριθεί στο, στα προγράμματα δράσης και αυτό αφορά και την αντίσταση στα μικρόβια. Τι έχετε κάνει με τα προγράμματα δράσης ως προς την αντιμετώπιση της ε, φυματίευσης και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού υφίστανται προβλήματα, ποιοι είναι οι τομείς όπου τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν το νομοθετικό πλαίσιο. Και αυτό αφορά και την Κομισιόν. Δεν μπορούμε να περνάμε στο επόμενο και στο μεθεπόμενο θέμα όταν δεν πληρούνται οι όροι για τα παρόντα προγράμματα. Εγώ θα πρέπει να φύγω να πάω σε άλλη συνεδρίαση, αλλά θα το παρακολουθήσω. Θα παρακολουθήσω την απάντησή σας κατά την αναμετάδοση. Ευχαριστούμε την κυρία Κονέτσνα. Ε, ο, ο κύριος Εικάουτ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερ για την παρουσία του. Θα ήθελα να μιλήσω για τους ε, ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς το αντιμετωπίζει η Επιτροπή. Το 2013 χρησιμοποίησε η Επιτροπή τη βέλτιστη νομοθεσία για να προωθεί σε μία μελέτη αντικτύπου ως προς τα επιστημονικά κριτήρια για τους διαταράκτες αυτούς. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ίδιο είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποφανθεί σωστά σε σχέση με τους επιστημονικούς δείκτες για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Δηλαδή, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της Κομισιόν. Υπήρχε μία αρχική πρόταση τον Ιούνιο του 2016, αλλά και τότε η Επιτροπή προσπάθησε να αλλάξει τον νόμο μέσα στα πλαίσια ε, μιας κατεξιοδότηση πράξης, μέσα στα πλαίσια του νομοθετήματος περί φυτοκτόνων. Έχουμε λοιπόν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και της βιομηχανίες, οι οποίες δεν θέλουν να δεχτούν ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Άρα η Επιτροπή θα προβάλλει επιστημονικά κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Το περιμένουμε χρόνια τώρα και το δικαστήριο αποφάνθηκε ένα μισή χρόνο πριν. Αλλά δεν θα πρέπει να αλλάξετε και το νομοθετικό κείμενο με μια κατεξουσιοδότηση πράξη όπως κάνατε στο παρελθόν. Δυστυχώς συμβαίνουν περίεργα πράγματα σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι εάν υπάρχει η καλύτερη γνωμοδότηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάτι τέτοια δεν πρέπει να συμβαίνει. Η κυρία Ντορνανό, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στην ανακοίνωση της 25ης Οκτωβρίου για το πρόγραμμα εργασίας για το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι θα δράσει υπέρ της κυκλικής οικονομίας και θα μειώσει το, τα πλαστικά και τη χρήση του στο περιβάλλον. Κατά την εφαρμογή του προγραμματός σας μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η, θέση του προγράμματος παραγωγής, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και ως προς την Αφρική και την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να προωθεί την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βελτιστοποιήσει τη συνεισφορά της ΚΑΠ στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς ε, το συμφιλιώνεται αυτό με το γεγονός ότι η ΚΑΠ έχει πρωταρχικό στόχο την αύξηση της ε, παραγωγικότητας με βάση το άρθρο 39 της ΛΕ. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, προστατεύοντας την ε, υγεία των ανθρώπων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς αντιμετωπίζουμε και τα παρασιτοκτόνα και τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς. Στον τομέα της ε, αεροπλαίας δεχόσαστε τον οργανισμό ΑΣΕΗ που θεωρεί ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αποφανθεί νομίμως επί του θέματος. Ευχαριστώ. Και έτσι τελειώνει ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τίμερμανς. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και αν δεν μπορώ θα σας απαντήσω αργότερα γραπτός ε, κάποιες ερωτήσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες οπότε ζήτησα από τους βοηθούς μου να δούμε αν μπορούμε να απαντήσουμε αμέσως αλλιώς θα απαντήσουμε γραπτός κάποια άλλη στιγμή. Κατάγει το θέμα της, των υπηρεσιών υγείας. Ήδη υφίσταται ένα νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα είναι ένα παράδειγμα. Ε, τώρα ο στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και να συνεχίσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή. Σε ό,τι αφορά τα θέματα υγείας, σύντομα ε, θα υιοθετήσουμε πρόγραμμα δράσης για την αντίσταση στα αντιβιωτικά και θα ενισχύσουμε τον αγώνα μας ε, εναντίον αυτού του φαινομένου, όπως ζήτησε ο κ. Λίζε. Επίσης, προετοιμάζουμε μια πρωτοβουλία για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, που θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. Ε, η εφαρμογή απαιτεί πολλή δουλειά ε, για παράδειγμα την οδηγία των πρώτων καπνού, ε, τις ε, διαμεθορικές υπηρεσίες υγείας και το νομοθετικό πρόγραμμα για τα φάρμακα. Όλα αυτά απαιτούν πάρα πολύ δουλειά από μας. Πολλά από αυτά που κάνουμε στηρίζουν τις πολιτικές των κρατών μελών, διότι όπως γνωρίζετε οι αρμοδιότητες μας είναι περιορισμένες. Εμείς χρησιμοποιούμε τι αρμοδιότητες που μας δίδονται για τα δημιουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων, ε, διάδοση βέλτιστων πρακτικών κλπ. Οπότε θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά που τους αναλογεί. Τώρα για τη γλυφοσάτη. Το συμπέρασμα της ΕΦΣΑ και της ΕΚΑ ότι η γλυφοσάτη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ε, καρκινογεγόνος ε, νομίζω ότι ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα και άλλων ρυθμιστικών φορέων εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών Καναδά, Αυστραλίας, Νέα Ζηλανδία Ιαπωνίας και του, ε, του κοινού φόρουμ του ΟΗΕ. Το μόνο αντίθετο στοιχείο που έχουμε, μάλλον το μόνο στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μα είναι οι επιστημονικές ένδειξεις ε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα συναισθήματα ε, ή σε οποιαδήποτε πολιτικά επιχειρήματα ε, να θέσουν στο περιθώριο τις, τα επιστημονικά πορίσματα. Στις 16 Μαΐου το Κολέγιο των Επιτρόπων συμφώνησε ότι θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας της για 10 χρόνια λαμβάνοντα υπόψη τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τα συμπεράσματα τα οποία μόλι σα ανέφερα. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να βρούμε μια λύση που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη και προφανώ το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασία τη ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλοντο, όπω προβλέπεται από την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμενη στα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία και ε, στον νόμο. Κύριε Έκτχαουτ, θα πρέπει να βασιστούμε στον νόμο. Ε, η προθεσμία για την ανανέωση είναι έξι μήνες μετά την αύξηση της ε, αίτησης. Η γνωμοδότησή μας θα είναι έτοιμη κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Τα κράτη -μέλη, ε, η συζήτηση με τα κράτη-μέλη θα γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το φθινόπωρο θα γίνει η ψηφοφορία για την στρατηγική βιοπικιλότητας το πρόγραμμα δράσης Natura και το συζήτησα και την περασμένη εβδομάδα επί Μακρόν με τους ε, εκπροσώπους ε, των ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών να ανησυχούν για τη βιοπικιλότητα. Αυτές οι ανησυχίες υφίστανται παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτές τις ανησυχίες και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και μάλιστα στο πρόγραμμα δράση που υποβάλαμε την περασμένη εβδομάδα είναι φανερά αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε, αλλά ε, είναι προφανέ ότι τοπικέ κοινωνίε ακόμα δεν βλέπουν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λόγο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Ε, το περιβαλλοντικό dumping είναι πράγματι ζήτημα ως συνέπεια πολιτικών επιλογών που δυστυχώς δεν έχουν μόνο, σχέση, δεν έχουν μόνο σχέση με, αυτούς, με αυτές τις χώρες που έχουν επιλέξει να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις υπόλοιπες. Σε πολλά κράτη-μέλη ε, θεωρείται ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα και η νομοθεσία ε, είναι, προέρχεται από αόρατους και γκρίζους υπαλλήλους στην ε, Βρυξέλλες παρόλο που οι δικοί τους εκπρόσωποι στο Συμβούλιο τα έχουν ψηφίσει. ε, ε υπάρχει το επιχείρημα ότι το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ κάνει καλό στην οικονομία αλλά αυτό είναι πραγματικά ξεπερνάει και τα όρια της ηλικιότητας. Ε, είναι ψευδές ότι ε, υφίσταται μια τέτοια πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν η οικονομία μας να αυξάνει το βάρος στο περιβάλλον. Το, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο μελλοντικά. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε ότι η οικονομία μας θα πρέπει να βοηθάει στο να μειωθεί το βάρος προς το περιβάλλον και οι πολιτικές μας το λέω ως εγγονός δύο ανθρακορίχων, οι πολιτικές αναζωπήρωσης της παραγωγής άνθρακα δεν κατανοούν ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες πηγές ενέργειας και άλλες δουλειές για τους ανθρακορίχους. Ε, ε, δεν θα πρέπει να χειροτερεύσουμε την ζωή των ανθρακορίχων και των κοινωτήτων αυτών. Ε, εγώ γνωρίζω πόσο οδυνηρή είναι η ζωή των ανθρακορίχων. Ξέρω πόσο δυνηρές ήταν ε, στο παρελθόν οι μεταρρυθμίσεις, αλλά ε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των άλλων πηγών ενέργειας. Ε, κύριε Κονέτσνα, με ρωτήσετε την εφαρμογή. Θέλω να σας καθυσυχάσω Έχουμε υποχρέωση ως θεματοφύλακες των συνθήκων να αναγκάζουμε τα κράτη-μέλη να σέβονται την νομοθεσία, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και η Κομισιόν θα αποδείξει ότι θα, ε, αν χρειαστεί θα ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάση αν αυτή είναι η μοναδική οδός που θα μας έχει απομείνει. Γιατί, γιατί επιμένω πως πρόκειται για το μέλλον μας, δεν πρόκειται για μια πολυτέλεια. Κάθε οικονομικό μοντέλο, οποιοδήποτε οικονομικό μοντέλο βιώσιμο για το μέλλον μπορούμε να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε, έχει ως κομμάτι την ε, εφαρμογή της ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, να σας προσπαθήσω να απαντήσω ότι στην λεπτομερή σας ερώτηση, κύριε Κάουτ, ε, δεν μπορώ να σας δώσω μια πλήρη απάντηση σήμερα, λυπάμαι. Δεν έχω αυτές τις προφορίες μαζί μου σήμερα. Ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και ε, θέλουμε να ε, υιοθετούν κριτήρια. Επειδή ήσασταν πάρα πολύ σαφείς όμως, δεν θέλω να σας δώσω μια πρόχειρη απάντηση. Θα σας δώσω μια γραπτή λεπτομερή απάντηση, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Αντωνάνο, και εσείς είχατε μια πολύ, μάλλον κάποιες πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις. για το ε, θέμα ε, της, της βραχικυκλώματος, ε, δηλαδή ε, το πώς τόπου μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και μείωση των τοπικών αποβλήτων. Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που βλέπουμε. Για παράδειγμα, η παροχή ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων, όλα αυτά γίνονται πιο προσωπικά, πιο ατομικά, πιο τοπικά και είναι σημαντικό οι τοπικές κοινωνίες να εμπλακούν. Ε, προφανώς ο σχεδιασμός θα είναι συνολικός, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι τοπικές κοινωνίες να εμπλέκονται. Το ίδιο και για τον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε τους στόχους για τη βιοποικιλότητα, να εξασφαλίσουμε βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, να εξασφαλίσουμε την διατήρηση του περιβάλλοντος μας χωρίς πλήρη συμμετοχή του αγροτικού πληθυσμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και σίγουρα δεν είναι δυνατόν ε, να κάνουμε οτιδήποτε ενάντια στη βούληση των αγροτών. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σε συνεργασία. Δηλαδή ε, το να καταστήσουμε πιο οικολογική την γεωργική παραγωγή απαιτεί τη συμμετοχή των αγροτών. Και πολύ σωστά αναφερθήκατε στη συνθήκη σε ό,τι αφορά τον στόχο της κοινή αγροτικής πολιτικής. Αυτός ο στόχος όμως όπως αναφέρει τη συνθήκη, θα πρέπει να εφαρμοστεί με, σήμερα με τρόπο διαφορετικό από ό,τι πριν από 15 χρόνια. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Χρειάζεται να θρέψουμε περισσότερους ανθρώπους και μάλιστα με έναν τρόπο πιο βιώσιμο. Έτσι ώστε ε, η, η φύση μας ε, να μην αποδεκατιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων τους Ευρωπαίους και με τρόπο περιβαλλοντικά ε, βιώσιμο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν καταλαβαίνω πώς η μετανάστευση συνδέεται με αυτά που είπατε. Αλλά να σας πω τη δική μου άποψη προσωπική. Ένα μεγάλο κομμάτι της μετανάστευσης ε, προκύπτει, είναι αποτέλεσμα ερημοποίησης, κλιματικής αλλαγής, ε, περιβαλλοντικών προβλημάτων κλπ. Η, τα επιστημονικά στοιχεία είναι τόσο απόλυτα ότι η μετανάστευση, ή ε, μάλλον ότι ε, οι αλλαγές στο περιβάλλον προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα που ε, πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στην Αφρική Διατήρηση διατήρησης της ε, διατήρηση και αύξηση των υδάτινων πόρων κλπ. Συνδέεται το περιβάλλον με τη μετανάστευση ασφαλώς σκεφτείτε η, τη λειψιδρία. Πώς έχει επηρεάσει αυτό τις αυτή τις μεταναστευτικές ροές. Και προφανώς έχει οδηγήσει και σε μεγάλο αριθμό ε, ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να ε, περάσουν, διασχίσουν την Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά τα καταφέρατε. Νομίζω απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν ε, είναι ικανοποιημένοι οι ερωτήσαντες, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον ό,τι αναφέρθηκε το σχολιάσατε. Τώρα θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωταπαντήσεων με άλλους συναδέλφους ε, και με πρώτο τον κύριο Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, Παρίσι. Συμφωνία των Παρισίων μετά από όσα συνέβησαν στη Βόσιγκτον. δεν έχει απλά αποσυρθεί ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές, αλλά υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για το πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο μέλλον. Μεγαλύτερη ανησυχία. Ε, ακούστηκαν πολλά τις τελευταίες ημέρες και θα μπορούσε να είναι ε, εύκολο να υποκύψουμε σε αυτόν τον ε, πειρασμό, να έχουμε αυτό το φόρο εισαγωγής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλή ιδέα. Το θέμα είναι άλλα εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τις χώρες που δεν σέβονται τις δεσμεύσεις τους ε, στο πλαίσιο της συμφωνίας. Να τα περιλάβουμε στο σύστημα ETS. Ε, είπατε και στην ε, αρχική σας παρέμβαση ότι διαπραγματευόμαστε τη μεταρρύθμιση του ETS. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Financial Times έγραψαν ότι οι μηχανισμοί που θα καλύπτουν τις αγωγές θα μπορούσαν να είναι πολύπλοκοι, άκρος πολύπλοκοι. Η Καλιφόρνια όμως δεν κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Το Φεβρουάριο ετέθη, επιτάπτωση πριν από κάποιους μήνες, στην πρόταση μεταρρύθμισης ε, για το πρόγραμμα ανταλλαγής ε, για το πολιτεία της Καλιφόρνιας. Αν λοιπόν οι εισαγωγέ από τη ΣΥΠΑ εντάσσονται από την Καλιφόρνια στο δικό της το σύστημα που είναι παρόνιο με το Ευρωπαϊκό, μήπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε και αυτή να βρει μια νομική ανθεκτική λύση νομικά ευσταθή δηλαδή και λογική λύση. Να συνδέσουμε ίσως το σύστημά μας με την Καλιφόρνια, με το σύστημα της Νότιας Κορέας και άλλα συστήματα που ισχύουν σε παγκόσμιο σε άλλες χώρες για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Και τις εταιρείε που θέλουν να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τις εντάξουμε κατά την ίδια γενική κατηγορία. Πρώτος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλετ που αναφερθήκατε στο ETS. Κύριο Σπαρνιά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω και εγώ στην αποχώρηση του Τραμπ από την COP21. Πολλοί παρατηρητέ σήμερα λένε ότι θα εφαρμοστεί χωρί τον Ντόναλτ Τραμπ η συμφωνία, αλλά όχι χωρί τη ΣΥΠΑ. Και ο Αμερικανικό λαό, το βλέπουμε τι τελευταίε εβδομάδε, δεν είναι έτοιμο να ακολουθήσει τον νέο του πρόεδρο. Μετά την ανακοίνωση απόσυρσης, ε, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει ένα μέτωπο κατά του Τραμπ για το κλίμα. Ιωνίου. ο Μάικλ Μπλουμγκαρ, τέος δήμαρχος ε, της Νέας έχει ε, στείλει μια υποστα... επιστολή στον ΟΗΕ που την υπογράφουν χίλιες οργανώσεις από τη ΣΥΠΑ που λένε ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε κατά 20% με το 2025 τις εκπομπές που ήταν ε, και η δέσμευση του Ομπάμα στην COP21. Λέει δηλαδή είμαστε ακόμα μαζί σας αυτή η επιστολή. Επίσης, περιφερειακές τοπικές ε, οργανώσεις τελικά έχουν πολύ περισσότερο βάρος ε, και αρμοδιότητες από τις κυβερνήσεις ό,τι αφορά την καταπολέμηση ατμοσφαιρικής ε, ρήπανσης και την εφαρμογή νέων περιβαλλοντικών κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει, κατά την άποψή μου, πολύ γρήγορα να ξεκινήσει συνεργασία σε τρία επίπεδα με τις Αμερικανικές πολιτείες, τις πόλεις και τις επιχειρήσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε, λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε, εσείς έχετε μια ατζέντα πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού θα μπορούσε να ενισχύσει τις σχέσεις της ε, με τις πολιτείες, με τους δήμους, με τις οργανώσεις, αμερικανικές επιχειρήσεις που είναι ευνοϊκές στο να ε, συνεχίσει η ΙΠΑ να εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Ομπάμα στην COP21. ευχαριστώ. Κύριος Λαβία τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, για την παρουσία σας σήμερα και για τις λεπτομερείς απαντήσεις που μας δίνετε. Ως προς τη Συμφωνία των Παρισίων και την επιλογή του Τραμπ να αποσυρθεί, εμείς ενδιαφερόμαστε ε, για τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής που μάλλον θα είναι περιορισμένες. Τι θα κάνουμε όμως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβάλει ένα νομοθετικό πακέτο για την κυκλική οικονομία, το ETS, ε, το Λούλους και ε, τον επιμερισμό προσπαθειών. Υπάρχει όμως και ένα νέο πρόγραμμα της Επιτροπής. Τι θα κάνει ακριβώς για τη διαδικασία εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων. Πώς θα κινηθεί η Κομισιόν κατά το επόμενο πρόγραμμα εργασίας επί του θέματος. Γιατί θέλουμε έγκαιρες πληροφορίες επί του θέματος για να μπορέσουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσουμε ορισμένες υποδείξεις πριν υποβληθεί η τελική πρόταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ στη Συμφωνία των Παρισίων, που είναι ένα θέμα που μας θίγει άμεσα. Θα ήθελα να προσθέσω όμως κάτι σε σχέση με τους προλαλήσοντες. Αυτή η απόφαση είναι οριστική από πλευράς, είπα από ό,τι φαίνεται. Και στην Ιταλία, στη Μπολόνια, επιβεβαίωσαν αυτή την απόφαση, απόφαση συγγνώμη, ε, ως απόρρια των G7. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο. Γιατί πέρα από την πρόκληση αυτή θα πρέπει να έχουμε χαμηλή χρήση άνθρακα και υπάρχουν και πολλές προκλήσεις στον τεχνολογικό τομέα. Γιατί όποιος εφαρμόζει αυτό το πλαίσιο θα είναι και πιο ανταγωνιστικός. Αλλά για να είμαστε αξιόπιστη δεν θα πρέπει μόνο να προβάλλουμε στόχους, αλλά να φτάσουμε σε αυτούς και εσείς ως ε, πραγματιστής γνωρίζετε ότι φτάνουμε στους στόχους μόνο όταν κάνουμε επενδύσεις. Άρα χρειάζεται ειδική γραμμή του προϋπολογισμού. Ε, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και το σύμφωνο σταθερότητας και ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της ε, βιώσιμης κινητικότητας και της ε, κυκλικής οικονομίας. Ποια είναι η άποψή σας επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαχαβωνή. Ε, έκπληξη, έκπληξη για μένα αποτέλεσε ε, ε, απετέλεσαν τα ε, λεγόμενά σας και το θέμα που επιλέξατε. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις, τις οποίες θα διατυπώσω στα ουγγρικά. Όταν εξελέγει ο πρόεδρος Γιούνκερ, αναφέρθηκε σε διάφορα περίπλοκα θέματα και τώρα θα πρέπει να αποφασίσει για την ντουπόν, την Μονσάντο, τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και ιδιαίτερα το καλαμπόκι. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέριψε με μεγάλη πλειοψηφία την αδειοδότηση αυτών των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και δεν υποστήριξε το Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την αντίσταση των κρατών μελών καθίσταται σαφές ότι στην Ευρώπη δεν θέλουμε να επιτρέψουμε τα προϊόντα αυτά, τους γενετικώς τροποποιημένους αυτούς οργανισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα διαχειριστείτε αυτό το θέμα. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε ε, εδώ μαζί μας. Δεν ήμουν εξ αρχής εδώ, αλλά μας, μου είπανε ότι είπατε πολλά για τους ε, βιώσιμους στόχους της χιλιετίας. Έχουν γίνει πολλές συστάσεις της Επιτροπής ε, που μας βρίσκουν σύμφωνους. Και ως προς το πολυεταιρικό φόρουμ, μάλλον τον φόρουμ των ε, εμπλεκομένων φορέων, θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο θα γίνει μία συζήτηση σε επίπεδο τοπικών και εθνικών αρχών καθώς και ευρωπαϊκών. Μπορείτε να μας πείτε αυτά παραδείγματα για το πώς βλέπετε τη λειτουργία αυτού του φόρουμ. Ο κύριος Φλόρενς. Ευχαριστώ πολύ. Για τον κύριο Τράμπα. Πραγματικά είναι ένας αγιατολά ε, του κλίματος. Ε, δεν θα τον φοβόμουν και πολύ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της κλιματικής πολιτικής πραγματικά εργαστεί κοινοτόμα και αν είναι καινοτόμα ε, η βιομηχανία δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει η αμερικανική βιομηχανία την ευρωπαϊκή βιομηχανία αν θέλει να κρατήσει πρωτεία ε, στην παγκόσμια αγορά. Δηλαδή ε, σίγουρα δεν είναι ο Τραμπ ε, ένας ε, φίλος, αλλά νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθήσουμε τη δική μας ε, πολιτικές. Σε ό,τι αφορά άλλα θέματα, κύριε Αντιπρόεδρε, μου άρεσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας σας. Αναφέρατε 17 τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά αφήσατε κάπως ανοιχτή την αλυσίδα, γιατί υπάρχουν κάποια κενά Κάποιοι κρίκοι λείπουν. Θα ήθελα λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί και να μην κατάλαβα καλά, να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, σε ό,τι αφορά το clean air, είναι πολύ σημαντικό. Ε, ένα σχέδιο δράση ε, που είπατε, τι περιλαμβάνει. Εγώ λαμβάνω πολλές καταγγελίες από φορείς στη χώρα μου και ως αγρότης με ενδιαφέρει σίγουρα και το θέμα της φυτοπροστασίας. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια νέα γενιά αυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα νεονικοτινοειδή. Καλό θα ήταν να απαγορευθούν άμεσα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στη βιομηχανία ότι ε, χρειάζεται μια νέα γενιά αυτοπροστατευτικών ε, ε, προϊόντων. Αλλά με ενδιαφέρει και το θέμα της ε, προστασίας ε, του νερού, του υδροφόρου ρίζοντα. Χρειαζόμαστε νέα μέσα ε, και αυτή η επιμήκυνση, αυτή η καθυστέρηση συνεχώς και αυτό πραγματικά είναι καταστροφή. Χρειάζεται μια νέα γενιά. Αν μπορείτε λοιπόν να μας πείτε δύο-τρία πράγματα και βέβαια για τα γεωργικά θέματα. Σίγουρα έχω να πω πολλά, γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα ε, συνείδησης, πώς να το πω, και εμείς και οι συνάδελφοι ε, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική βιωσιμότητα, ε, πρέπει να αλλάξει η αντίληψη γενικώ, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση για τους νέου αγρότες ε, καλύτερα είναι τα πράγματα, αλλά η νοοτροπία των αγροτών τη δική μου ηλικία είναι καταστροφική. Θα πρέπει να τους εξηγήσουμε λοιπόν πού πηγαίνουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας για να τους έχουμε στο πλευρό μα. δεν ε, βοηθάει τίποτα το να προσπαθήσουμε συναισθηματικά να επηρεάσουμε. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Εγώ έχω αρκετές ελπίδες. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τη σύμβαση του Άρχους. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης της ε, Σύμβασης του Άρχους στις 17 Μαρτίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβαίνει το άρθρο 9 της ε, σύμβασης αυτής. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την απονομή δικαιοσύνη δηλαδή. Καμία μη κυβερνητική οργάνωση δεν, ε, και κανένα άτομο δεν έχει λάβει την άδεια να ε, προβεί ε, ε, ε, να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιοδήποτε θέμα παράβασης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν του θέματος της μη αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων. Ε, η Επιτροπή Συμμόρφωσης του, της Σύμβασης του Άρχους ε, κατέληξε αυτό το συμπέρασμα και τα συμπεράσματά της πάντοτε από το 2002 τα λάβαναν υπόψη και τα δέχονταν τα κράτη-μέλη στην Συμφωνία των Μερών με την ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, για αυτό το συμπέρασμα της Επιτροπής Συμμόρφωσης, τι θα πράξει η Κομισιόν, δεδομένου ότι βρίσκεται στο εδόλιο. Ευχαριστούμε κύριε Ένα από τα θέματα ε, είναι η Λούλουσεφ ε, για τη χρήση γης και τις αλλαγές χρήσης γης. Ε, υπάρχουν δύο θέματα στα οποία συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες, παρόλο που υπάρχουν άλλες διαφωνίες. Πρώτον, ότι θα πρέπει να φυτέψουν περισσότερα δέντρα, γιατί απορροφούν ε, διοξείδιο του άνθρακα. Και δεύτερον, θα πρέπει να αυξήσουμε την οικοδόμηση σε ξύλο, κατασκευή ακίνητος ξύλινων ακινήτων. Γιατί ε, αντικαθίσταται το τσιμέντο, ε, μιλήσατε για τα πλαστικά και πόσο σημαντικά είναι ε, στην μόνη του περιβάλλοντος, αλλά ε, το 8% των εκπομπών άνθρακα παγκοσμίω οφείλεται στη τσιμεντοβιομηχανία. Οπότε καλό είναι το τσιμέντο να το αντικαθιστούμε με ξύλο. κάτι που όμως εμποδίζει την αύξηση της χρήσης του ξύλου στα ακίνητα ε, είναι οι κανονισμοί για την πυρασφάλεια. Η άφηξη ε, καινούριων ξύλων προϊόντων ε, ε, που προστατεύουν εξωτερικά τα, τις οικοδομές μπορεί να ε, βελτιώσουν την κατάσταση διότι επιτρέπουν σε ένα φλεγόμενο κτίριο να γνωρίζουμε πότε θα καταρρεύσει ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με, τα, ε, με το τσιμέντο και τον πετόν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε για ανηγενίασαν το πρώτο 12όρφο ξύλινο κτίριο στο Portland και στην Βιέννη του χρόνου ένα παρόμοιο κτίριο θα έχει 24 ορόφους. Βλέπουμε λοιπόν σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με την χρήση ξύλινων κτηρίων. Εσείς ε, θα επωφεληθείτε της ευκαιρίας, των ευκαιριών που θα παρουσιαστούν μπροστά σας για να στηρίξετε αυτή την τάση. Άλλοι συνάδελφοι, αν έχουν ερωτήματα, να τα δείξουν. Για να κλείσουμε τον κατάλογο ομιλητών. Ο Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Για μένα καθίσταται σαφές ότι πολλοί βουλευτές ε, έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη Συμφωνία των Παρισίων και τι ευθύνες αναλαμβάνουμε και πώς τις αναλαμβάνουμε έτσι ώστε να αποτελέσει επιτυχία παρά την απόσυρση του Προέδρου Τραμπ. Εκφράσαμε τη βαθιά μας απογοήτευση για την απόφαση αυτή, όμως μας ενθαρρύνουν τα πολλά σχόλια υποστήριξης εδώ από όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά και από πολλά ε, μέρη στις ΕΠΑ, στην New York Times είδα μία αγγελία όπου οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΕΠΑ υποστήριξαν ενεργά την ε, Συμφωνία των Παρισίων, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με βάση τα αμερικανικά συμφραζόμενα, ποτέ δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη όθηση για τη λειτουργία της Συμφωνίας των Παρισίων. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες, οι τοπικές αρχές και ούτω καθεξής γνωρίζουν ότι έχει αρχίσει η πλεύση αυτής της πορείας. Γι' αυτό συμφωνώ με σας που λέτε ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε και νέες ε, εταιρικές σχέσεις, δηλαδή όχι μόνο μεταξύ κρατικών οντοτήτων, γιατί να μην έχουμε καλύτερες ε, και πιο δυνατές εταιρικές σχέσεις έχνης με την Καλιφόρνια και υπάρχει η δυνατότητα ε, μιας κοινή πορείας μεταξύ Παρισίων και Πίτσμπουργκ. Η Συμφωνία των Παρισίων που από νομικής πλευράς δεν είναι η πλέον ισχυρή, είναι μία δήλωση προθέσεων από τον κόσμο, όμως θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για να αλλάξουν τα πράγματα ανά τον κόσμο, από πλευράς περιβάλλοντος και το καθεξής, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η προσέγγιση σύγκλησης κρατών μόνο σε κρατικό καθαρά επίπεδο. Και αυτό το βλέπω με εταίρους που θέλουν ε, επαφές μαζί μας, όχι μόνο τους ε, Κινέζους. Θέλουν δηλαδή να αναλάβουμε αυτό τον ηγετικό ρόλο. Το επιθυμούν για να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική πορεία. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουν οι λαοί μας κατά πλειοψηφία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κύριος Μπέλετ αναφέρθηκε σε αυτό, καθώς και άλλοι. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε τον άνθρακα. Δηλαδή να ξέρουμε ποιο είναι το κόστος του, να μην μιλάμε μόνο για μια πολιτική τιμολόγησης καθαρά, αλλά την πίεση που θέτουμε ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος ε, ανταλλαγών εκπομπών. Έχει γίνει πολύ και σημαντική εργασία μεταξύ των συνομοθετών επί του θέματος, αλλά τώρα χρειαζόμαστε την πολιτική θέληση για να δώσουμε μία όθηση στις διαπραγματεύσεις και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια από τη δική μου πλευρά να μιλήσω με τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων γιατί έτσι μπορούμε μόνο να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας ότι είμαστε πολύ σοβαροί και θέλουμε το δικό μας ETS να ανταποκριθεί στους στόχους των Παρισίων. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να επιτευχθεί. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε μέτρα ε, σε σχέση με τα σύνορά μας. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε γιατί και ο ΠΟΕ θα μας ε, κατηγορήσει γι' αυτό εάν το κάνουμε. Δεν ξέρω καν αν είναι και ευκταίο δεν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη ούτε οι εμπλεκόμενοι φορείς. Γι' αυτό νομίζω ότι το δικό μας σύστημα ανταλλαγής εκπομπών μας οδηγεί σε ένα σύστημα επιμερισμού στα κράτη-μέλη και διατομεακά. Διαφορετικά χάνουμε τη δύναμή μας. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξο επ' αυτού. Ο κύριος Λαβία μας ρώτησε τι σημαίνει αυτό για την εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τη δική μας πλευρά. Το μήνυμά σας ε, ελήφθη και θα δω τι μπορούμε να κάνουμε για τον επόμενο χρόνο και τις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό σχετίζεται και με τις επενδύσεις Είχαμε μια διάσκεψη στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ ε, βρέθηκα στη Νέα Υόρκη εδώ και τέσσερις εβδομάδες για να μιλήσω με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος για επενδύσεις, αλλά θα ήθελε νομική ασφάλεια από εμάς μακροχρόνια. Αυτή είναι η προαπέτηση των επιχειρήσεων για μακροχρόνιες επενδύσεις θέλουν μια νομική ασφάλεια μέχρι το 2030. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα. Ο ορίζοντας 2020 δεν είναι επαρκής για τον ιδιωτικό τομέα, για επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε επιτυχείς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ορίζοντα 2030 και φυσικά να συμβαδίσουμε με τους στόχους μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ίδια όθηση όπως έγινε τότε υπό τον Τελόρ το 1992. Πρόκειται για ένα πολύ δαπανηρό εγχείρημα. Και φυσικά όλοι θέλησαν να ενταχθούν σε αυτήν την αγορά και είχαν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Άρα, αν λάβουμε υπόψη τον ορίζοντα 2030, τότε θα, μπορέσαμε να αρκεστούμε, θα μπορέσουμε να αρκεστούμε στους παγκόσμιους στόχους και στο, στα πλαίσια ενός επενδυτικού προγράμματος. Σε σχέση με το φόρουμ αυτό, ε, το, φόρουμ όλων των εμπλεκομένων φορέων, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να είναι διαλειτουργικό. Και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη τις ε, τοπικές και εθνικές αρχές που αποζητούν στενή συνεργασία με την ε, Επιτροπή των Περιφερειών και όπου προβάλλεται μία συνεργασία στον τοπικό και περιφερειακό τομέα. Άρα προσπαθούμε να αποκεντρωθούμε κάπως από τις Βρυξέλλες μέσω αυτού του, του φόρουμ. Η Επιτροπή των Περιφερειών κατανοεί ότι θα πρέπει να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός έτσι ώστε αυτή η πλατφόρμα να κινηθεί λίγο εκτός ε, ε, ξελών. Και θα υπάρχει και μία διαχειριστική επιτροπή που θα διοργανώσει διάφορες δραστηριότητες και θα ε, αποδίδει, θα κάνει μάλλον μία έναν απολογισμό δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε μάλλον κάτι το οποίο να δείχνει πώς εργαζόμαστε. Κατανοώ τα σχόλια του κυρίου Φλόρενς για τους αγρότες. Απάντησα σε μια προγενέστερη ερώτηση, αλλά για να είμαι απόλυτα σαφής, θα ήθελα να πω ότι δεν θα φτάσουμε στα ποθητά αποτελέσματα χωρίς τους αγρότες ή κινούμενοι κατά των αγροτών. Θα πρέπει να έχουμε τη συμμετοχή τους. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και νέες τεχνολογίες για να βοηθήσουμε τους αγρότες να ενδώσουν. Ιδιαίτερα στο θέμα της πράσινης οικονομίας, το οποίο δημιουργεί διχασμούς. Εκεί που υπάρχουν μεγάλες γεωργικές, μάλλον, συγγνώμη, μικρές γεωργικές ε, εκμεταλλεύσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους αγρότες να ανταποκριθούν. Γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες τηλεδιαχείρισης, και διαλειτουργικότητας συστημάτων. Όταν μιλάτε με νέους αγρότες βλέπετε ότι δεν, δεν μπορούν να παραναδεχτούν αυτές τις ε, τεχνολογικές απαιτήσει και προκλήσεις. Έτσι θα μπορέσουμε να καταρρύψουμε και στερεότυπα που υπάρχουν σε αυτό το τομέα. και να έχουμε διαφορετικά σημεία κίνησης. Ως προς τη σύμβαση του Άρχους, κατανοώ το πρόβλημα που έθεσε η κυρία Χάρμς, προσπαθούμε να ορίσουμε τη θέση μας και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να κατανοούμε τη νομική μας θέση κατά την προσχώρηση στη Συμφωνία του Άρχους είχαμε πει ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι ε, ένομες σχετικά με το δικό μας δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο. Θα πρέπει δηλαδή να συμβαδίζουν με το κοινοτικό δίκαιο και την κοινοτική ένομη τάξη. Γι' αυτό ε, όπως είπε και η κυρία Χάρμς, εδώ υπάρχει ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και φυσικά δεν μπορώ να προχωρήσω πιο πέρα γιατί θα πρέπει να υπάρξει μία αποσαφήνιση του πλαισίου σε σχέση με τη χρήση των υγεών και τη δασοκομεία. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ε, θα ήθελα να σταθώ στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Θα σας μιλήσω προσωπικά, γιατί έχω κάποια πείρα επί του θέματος. Και τώρα, αλλά και όταν ήμουν υπουργός και το συζητούσαμε στο Συμβούλιο, τότε για μένα ως υπουργό ήταν πολύ δύσκολο να δούμε το πλαίσιο αυτό ολιστικά. Δηλαδή μόνο ε, ένα κράτο μέλος είχε αντιταχθεί, αλλά για λόγους επιτροπολογίας δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί οι κανόνες επιτροπολογίας ορίζουν ένα διαφορετικό πλαίσιο. Και γι' αυτό δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική η κατάσταση, γιατί δεν την κατανοούσε και η κοινή γνώμη αλλά ήταν τελεστικό και για τα κράτη-μέλη να πούνε ναι, προσπαθήσαμε να το σταματήσουμε, να σταματήσουμε αυτό το πλαίσιο, αλλά δεν με επέτρεψε η Κομισιόν να κινηθούμε περαιτέρω. Και η γλυφοσάτη λοιπόν είναι κάτι το οποίο ενοχλεί ακόμα και τον Ζαν Κλοντ Ιούνκερ. Γίνεται μια πολιτική συζήτηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται με βάση τους κανόνες της επιτροπολογίας. Θα πρέπει να αποφανθεί δηλαδή η Επιτροπή και στο τέλος τα κράτη-μέλη τι κάνουν. Λένε «Α, εμείς πολύ το θέλαμε, αλλά τελικά αποφάνθηκε διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Θα πρέπει όμως και οι πολιτικοί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και όχι να απεκδίονται των ευθυνών τους. Έτσι το βλέπω εγώ προσωπικά. Νομίζω ότι το μόνο μας όριο είναι οι επιστημονικές αποδείξεις. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν διπλό και τριπλό έλεγχη, αλλά εάν υπάρχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να τα δεχτούμε και ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει την πολιτική του ευθύνη και στο Συμβούλιο. Σε σχέση με τη χρήση των γεών και τη δασοκομεία, δεν ήξερα γι' αυτό το κτίριο το οποίο προαναφέρεται που έχει χτιστεί από ξύλο. Έτσι ίσως μπορεί να αλλάξουμε τον τρόπο που ε, χτίζουμε, πώς βλέπουμε και πώς αντιμετωπίζουμε το τσιμέντο. Τα τελευταία 15 χρόνια έχω έχω δει ε, τη μεγαλύτερη χρήση του τσιμέντου σε σχέση με 3.000 χρόνια πριν. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ανακύκλωση υλικών κατά την οικοδόμηση και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δασοκομεία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και βιωσιμότητα στα δάση. Αυτό αποτελεί και μέρος της ατζέντα για τη βιοπικιλότητα. Εάν είναι μονοδιάστατη η δασοκομεία, δεν θα μας ικανοποιήσει. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνεκτική στρατηγική. Και επί αυτού του θέματος σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προσπάθησα να απαντήσω στις ερωτήσεις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν ε, δεν είσαστε ικανοποιημένοι θα ήθελα να αποτανθείτε σε μένα και στους συναδέλφους γιατί ίσως δεν είχα όλα τα στοιχεία που επιθυμούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, περιμένουμε μια ηγετική στάση της ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά την αξιοπιτυχιστία των στοιχείων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανισμών. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν συζητά την αλλαγή της μεθόδου εργασίας της ΕΚΑ έτσι ώστε να μην εξαρτάται από εκθέσει των κρατών μελών, από στοιχεία των κρατών μελών, αλλά να προβαίνει σε ειδικέ τη ε, μελέτε. Ίσως κάτι τέτοιο θα έπρεπε να το σκεφτούμε, όχι αυτή τη στιγμή βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ και για την ε, προσωπική σας ε, εμπειρία, την, προσωπικέ σα σας αναμνήσεις σε ό,τι αφορά τον άνθρακα και τους ανθρακορίχους. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή τύχη. Dear colleagues, uh, this... Uh, εδώ τελειώνουμε τη συνάντησή μας για σήμερα. Επόμενες... Ε, όχι. Ε, η πρόταση της ε, Δημοκρατίας των ε, Νίσων Μάρσαλ θα είναι στο Κοινοβούλιο την Τετάρτη. Επόμενη συνεδρία στις 21, επόμενη συνεδρία στις 21 Ιουνίου. Ευχαριστώ.